Ανανεώνεται Präsident. Ανανεώνει τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα πρακτικά της χθεσινής ε, συνεδρίασης και τα εγκεκριμένα κείμενα είναι διαθέσιμα. Έχετε αντιρρήσεις σχετικά. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά λοιπόν. Επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης είναι η ερώτηση προς την Κομισιόν.